απελευθέρωση της έδρας του. από την 7η Οκτωβρίου 2009. Από την διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων έλαβα πρόταση για τον διορισμό των μελών της έκτακτης ε, επιτροπής για ε, την οικονομική κρίση. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα και θα, δια... θα ε, δημοσιευθούν και, στην... και στα πρακτικά. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών έχει οριστεί μέχρι αύριο 5η στις 9 η ώρα. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει στις 11 πάντα αύριο. Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε στην ε, έκθεση της κυρίας Ρενάτε Βέμπερ για την ε, πρόληψη και τον διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικέ